έτοιμα για να διορίσει τον κύριο Πασκάλα Ριμό ε, στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και τη Βαρόνη Νοσίνα Μομπαρίκ στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε αντικατάσταση του κυρίου Τζον Φλακ. Υπάρχουν μήπως αντιρρήσεις για τους δύο διορισμούς? Όχι, οπότε εγκρίνονται. Περνάμε στο επόμενο θέμα στη Μιανμάρ και ιδίως στην κατάσταση των Ροχίνγκια στη χώρα αυτή. Έχουμε έξι συντάκτες ε, του ψηφίσματος. Η πρώτη είναι η κυρία Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξάρσεις βίας στη Μιανμάρ που είναι σαν να προέρχονται από ένα βιβλίο ε, οδηγιών, ένα εγχειρίδιο γενοκτονίας. Αυτά τα λέει η Επιτροπή Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Χρειάζεται να φτάσει εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα που δεν μπορούμε να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε. Αλλά η καταστολή του στρατού είναι βίαιη και ομή και δεν μπορεί να γίνει για αυτή παραδεκτή. Ε, είναι δυσανάλογη η βία που ασκεί ο στρατός και θα πρέπει οι αρχές να πάρουν τις αποστάσεις τους. Εμείς ζητούμε μια ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή εξεταστική που να μπορεί να μεταβεί και στην περιοχή. Χρειάζεται οπωσδήποτε βιώσιμη λύση το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει στους Ροχίνγκια είτε ηθαγένεια είτε ένα νόμιμο καθεστώς, ένα νομικό καθεστώς που να του προστατεύει και να του δίνει και δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι δραματική η κατάσταση των Ροχίνγκια και ε, περιγράφει πάρα πολύ καλά την ε, αντιδημοκρατική εκτροπή αυτή τη στιγμή στη Μιανμάρ. Είναι διπλός ο στόχος τους να εξαλείψουν μια εθνική μειονότητα αλλά και να καταστήλουν την ανεξιθρησκεία και την ελευθερία της θρησκείας καθότι πρόκειται για μουσουλμάνους. Για το λόγο αυτό η συμπεριφορά των αρχών της Βυρμανίας είναι ε, βαρύτατη, την καταδικάζουμε και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με το λαό της Μιαμάρ και τους Ροχίνγκια. Και επίσης ζητούμε από τον Μπαγκλαντές να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του και να μην κλείσει τα σύνορά του έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να ε, διέρχεται τα σύνορα. Εμείς υποστηρίξαμε την κυρία Αουν και τον αγώνα της για την ελευθερία τόσα χρόνια αλλά τώρα μας γυρίζει την πλάτη έθελο τυφλή ε, και μάλιστα ενθαρρύνει αυτές τις επιθέσεις. Αν εξακολουθήσει μπορεί το Κοινοβούλιο να αποφασίσει να της αφαιρέσει το βραβείο Σαχάροφ. Σας ευχαριστούμε κύριε Παντζέρη. Ο κύριος Γιουνού Αμαρτζή, παρακαλώ τώρα για ένα λεπτό επίσης. Ε, ένας ολόκληρος πληθυσμός ε, έχει καταστεί άπατρη χώρα, στην ίδια του την πατρίδα ε, και σιωπηρά αποδεκατίζεται. Η σιωπή σκοτώνει. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να δράσουμε κατανομάζοντας και στυλιτεύοντας τις θηριωδίες, να, κατα... να καταδικάσουμε τις απαγωγές, ε, τις διακρίσεις και τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος της ε, μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, που μάλιστα ενθαρρύνονται από τα υπερεθνικιστικά βιρμανικά κινήματα ε, και τις εκστρατείες που κάνει και τις επιχειρήσεις ο στρατός. Και μάλιστα θα πρέπει ε, να κατονομάσουμε τις ευθύνες τμήματος της κυβέρνησης και τις σας με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης της κυρίας Αν που ήταν και βραβευθείς με βραβείο Ζαχάροφ. Πραγματικά είναι ανάξια του βραβείου που τις είχαμε απονείμει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε αυτό το κοινό ψήφισμα στο οποίο καλούμε να τεθεί ένα τέρμα σε αυτές τις φαγές και τις θηριωδίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριο Μαρζή. Ο κύριος Μπασίρ έχει το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο Έρμαν Μπέρκ, αυτό που χρειάζεται η τυραννία είναι άνθρωποι που έχουν αγαθή συνείδηση απλώς να παραμείνουν σιωπηλοί. Και στο Μιανμάρ μερικοί θα, θα προτιμούσαν ακόμη και πιο στεναρό ε, ψήφισμα πιο αυστηρό. Άλλοι είπαν να περιμένουμε ακόμη ένα μήνα. Αλλά αυτή η κολυσιεργία και η χρονοτριβία επέτρεψε τι σφαγέ στη Ρουάντα και στη Στρεμπρένιτσα. Κάποιοι είπαν επίση ότι δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τις ε, ε, συνεχιζόμενες εμπορικέ μα διαπραγματεύσει με το Μιανμάρ. Πώ μπορούμε να σκεφτόμαστε εμεί το εμπόριο όταν τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν την ε, περίπτωση της Μιανμάρ ως ε, κλασικό παράδειγμα εθνοκάθαρση. Δεν μπορούμε να θέλω ότι φλούμε μπροστά στην τυραννία μόνο για εμπόρικού λόγου. και σίγουρα η τυραννία και η κατάσταση αυτή δεν θα πρέπει να είναι αντάλλαγμα για το εμπόριο. Και σίγουρα χρειάζεται μια αποφασιστική απόφαση και πυγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντω, πολύ φοβούμε ότι αν δεν εξετάσουμε όλοι πολύ σοβαρά ε, επιβολή κυρώσεων και διακοπή των εμπορικών συζητήσεων, δεν θα απομείνει ούτε ένας ροχίνγκια ζωντανό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ορμας Πάετ. Σας ευχαριστώ. Τα τελευταία στοιχεία για τους Ροχίνγκια που προσπαθούν να γλιτώσουν από την εθνοκάθαρση είναι συγκλονιστικά. Από ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια περίπου 400.000 ήδη έχουν περάσει τα σύνορα του Μπαγκλαντές. Παρά τις, την πολύ επικίνδυνη διαδρομή και τις ε, απάνθρωπες και αποτρόπες συνθήκες διαβίωσης των Μπαγκλαντές. Οπότε ή ε, θα πάνε στο, στον Μπαγκλαντές όλοι οι Ροχίνγκια ή θα έχουν πεθάνει μέχρι τον Οκτώβριο. Ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ρητά και κατηγορηματικά ότι αν οι θηριωδίες αυτές δεν σταματήσουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει κυρώσεις και συνέπειες ως προς τις ε, εμπορικές προτιμήσεις που απολαμβάνει η Μιανμάρ. Η απώλεια χρήσιμων επενδύσεων ίσως είναι το μόνο επιχείρημα που μπορεί να μεταπίσει τους ε, στρατηγούς της Μιανμάρ να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε για ιατρικές υπηρεσίες και ανθρωπιστική βοήθεια στους καταβλισμούς του Μπαγκλαντές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε μία μέρα ακόμη γιατί ήμασταν παρατηρητές αυτών των κτηνοδιών εδώ και αρκετό καιρό ήδη. Σας ευχαριστώ. Και τώρα κύριος Κρίστιαν Ντάν Πρέντα, τελευταίο συντάξη τη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι με θλίψη βλέπουμε την Αουν ε, Σανσουκή να εμφανίζεται ανίκανη να χειριστεί αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Τι επήγει τώρα, να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω θα πρέπει να επιμένουμε σε αυτό. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε να μην στείλει στην αντιπροσωπεία ίντα ε, μέλος της. Είναι αδιανόητο τώρα να πηγαίνει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στη Μιανμάρ αυτή τη στιγμή. Επίσης, η πρόταση που κάνουμε ως ομάδα του ΕΛΚ ε, την παρουσίασα πριν από λίγο, να στείλουμε ε, την Επιτροπή ΑΦΕΤ και την Επιτροπή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πάρα πολύ καλή προετοιμασία εκατέρωθεν των συνόρων και στη Μιανμάρ και στο Μπαγκλαντές. Όχι στην πρωτεύουσα, στα σύνορα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην πρωτεύουσα να ακούμε τις επίσημες δηλώσεις και ε, οι ομιλίες. Να ε, οργανωθεί σοβαρά και σωστά αυτή η αποστολή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι πολιτικές ομάδες και οι εκπρόσωποι τους. Πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Τσάμπα Σόγορ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό η δίωξη των Ροχίνγκια που είναι η μεγαλύτερη ομάδα ε, απάτριδα στον κόσμο δεν είναι νέο φαινόμενο. Ήταν στόχος δεκαετίες ολόκληρε και χιλιάδες έχουν χάσει τι ζωές τους. Αυτό που είναι διαφορετικό σήμερα είναι η ομότητα ε, του στρατού. Ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αναλογική με τις επιδρομές των ανταρτών. Πρόκειται για εθνοκάθαρση ε, υπάρχουν ε, σοβαρές ε, εκθέσεις που μιλούν για βιασμούς, για ακροτριασμούς γυναικών, για αποκεφαλισμούς παιδιών από το στρατό και για πυρπόληση των χωριών τους. Και όλα αυτά γίνονται σε μια διαδικασία που η Δύση θεωρεί εκδημοκρατισμό και όπου ο πρόεδρος είναι ε, μια κάτοχος ε, του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης ε, και κάνει όλες αυτές τις φαγές ο στρατός. Θα πρέπει εμείς οπωσδήποτε να αποφασίσουμε, να απαντήσουμε. Ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Σοράγια Πόστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κτηνοδίες και θηριωδίες ε, της Μιαμάρα δεν εντάσσονται στα δικά μας μοντέλα, ούτε καν στο βουδιστικό μοντέλο που είναι ειρηνικό. Σίγουρα έχει χάσει την έγκλη της, της ε, ηρωίδας, ε, της υπερμάχου της ειρήνης και της πολέμιου των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γιατί έμεινε σιωπηρή μπροστά σε αυτή την σφαγή. Είδαμε Όλος ο κόσμος έγινε μάρτυρας των σφαγών κατά της κοινότητας, ε, της μειονότητας Ροχίνγκια. Έχουμε ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, Ροχίνγκια που προσπαθούν να γλιτώσουν φεύγοντας προς τον Μπαγκλαντές και η κυρία Σανξουκή έμεινε σιωπηρή μέχρι τέλους και ο αγώνας της που κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε μάλλον επιστεγάστηκε με βραβείο Νόβελ Ειρήνης και με βραβείο Ζαχάροφ δυστυχώς ε, έχει απαξιωθεί. Θα πρέπει επιτέλους να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του Γκουεντζιέλ. το λόγο έχει ο Μιγγέλ Ουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ. Στη Μιανμάρ δεν έχουμε τεράστια εθνική και θρησκευτική δίωξη κατά το Ροχίνγκια, αλλά έχουμε και αναγκαστικές, αναγκαστικούς εκτοπισμούς ε, εκατοντάδων ακροτών για αρπαγή της γης τους. Ε, ο νέος νόμος ε, για τις απαλωτριώσεις επιτρέπει την εισαγωγή ξένου κεφαλαίου προ, προωθώντας βιομηχανίες. Έχουμε έτσι αρπαγή της γης και μονοπόλιο και του ύδατος. Και μάλιστα δεν έχουμε μόνο την τη σύγκρουση την εθνοτική και την θρησκευτική για τους Ροχίνγκια. Έχουμε και άλλα εμπορικά κριτήρια και μάλιστα πρόσφατα ε, ένα εκατομμύριο των Ροχίνγκια αφιερώθηκαν σε αγοροεπισητιστικά σχέδια από την κυβέρνηση της Μιαμάρ. Δεν μπορούμε να γίνουμε απλοί παρατηρητές αυτής της τραγωδίας. Θα πρέπει να στυλιτεύσουμε την παρενόχληση και την εκδίωξη αυτών των κοινοτήτων. Θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ της πράσπισης των γεών τους και της κοινότητας Ροχίνγκια και να ταχθούμε υπέρ των ακτιμώνων και των εκτοπιστέντων εξαιτία αυτής της ένοπλης σύραξης στην, στο Μιανμάρ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρέσπο. Περνάμε στη διαδικασία Catch Ο Χωσέ Γνάσιο Φαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, οι μουσουλμάνοι Ροχίνγκια που έχουν ε, χαρακτηριστεί ως ε, άπατρης ε, λαός και χωρίς φίλους είναι τα θύματα της αδιαφορίας του κόσμου και της καταπίεσης και της καταστολής. Είναι όμως πραγματικά δυσανάλογη αντίδραση στους αντάρτες των Ροχίνγκια αυτή η επίθεση του στρατού και Μάλιστα ε, αυτές οι θηρετήσεις προκάλεσαν την έξοδο 300.000 και προσφύγων προς τον Μπαγκλαντές. Είναι κατεπίγουσα η ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνεχίζονται οι κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οδηγούν σε θάνατο και απόγνωση ε, πολλών μελών τη Ροχίνγκη και εμποδίζουν τον εκδημοκρατισμό και την εθνική επανασυμφιλίωση και τι ελπίδε που είχαν δημιουργηθεί το 2015 με τη νέα κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί σε όλε αυτέ τι διώξει που έγιναν στην πολιτεία Ραχίν. Θα πρέπει να καλέσουμε την Αγκ Σαν Σουχίν, που είναι κρατικό σύμβουλο ε, του στη Μιανμάρ και μάλιστα ε, και βραβευθήσαμε ε, Νόμπελ Ειρήνη το 1990 και βραβευθήσε με το βραβείο Ζαχάροφ να αναλάβει τι ευθύνε απέναντι στις, στην θρησκευτική αυτή μειονότητα και να καταπολεμήσει οποιαδήποτε μορφή ριζοσπαστισμού. Δεν μπορεί να, να παραμείνει σιωπηρή μπροστά σε αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία. Ευχαριστώ. Ε, ε Η κυρία Τζολί Ward, παρακαλώ. Όλοι νιώθουμε τη φρίκη για τα όσα συμβαίνουν στους μουσουλμάνους Ροχίνγκια στην Μιανμάρ και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να εκφράσουν την ανησυχία τους. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μείνει ε, θεατής ενώ γίνεται μια ε, εθνοτική καθάριση ε, σύμφωνα με τους κανόνες όπως είπε και ο ΙΕ. Δεν, είναι αρκ... αρκεί το να το συζητάμε. Τέτοιε φρικαλαιότητε συνεχίζονται παρά τι δηλω... διπλωματικέ δηλώσει. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, χτίσει, να οικοδομήσει μια στεναρή στρατηγική για να αντιμετωπίζει τέτοιου είδου καταστάσει, για να ασκεί πραγματική πίεση ώστε να σταματήσει η βία και συνεργαστεί με του διεθνεί συνεργάτε και τι ε, οργανώσει κατά του ρατσισμού, ώστε οι δράστε να ε, φτάσουν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα της εθνικής μειονότητας στο Ροχίγια έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Ιούλιο του 2016, τον Δεκέμβριο του 2016 και βεβαίως στην ε, έναρξη τον Μάρτιο του 2017. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια εθνοκάθαρση και αυτό γίνεται καθαρά για οικονομικούς λόγους προκειμένου να γίνει αρπαγή της γης εκεί όπου κατοικούσαν οι κοινότητες των ροχίνγκια διότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για εξορίξεις ενδιαφέρον από μεγάλες πολυεθνικές. ταυτόχρονα αρπάζουν και την ε, εκμετάλλευση του ύδατος. επομένως η θρησκεία χρησιμοποιείται ως μια δικαιολογία. το ότι τυχαίνει οι ροχίγκια να είναι μουσουλμάνοι δεν έχει καμία σχέση διότι πίσω από όλα αυτά είναι μια διαδικασία οικονομική. αυτό πρέπει να δούμε και σε αυτό πρέπει να σταθούμε καταδικάζοντας τη βία από την πλευρά του στρατού και βεβαίως ζητώντας άμεσα μέτρα για να σταματήσει η εθνοκάθαρση η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη βυρμανία και θα περιμέναμε από την σου που έχει βραβευτεί και με το βραβείο ζαχάροφ να έχει πάρει μια θέση πολύ αποφασιστική. επομένως κυρία μογκερίνη περιμένουμε τη λήψη μέτρων από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, ε, Η κυρία ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Μογκερίνη. Τα είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Οι εκθέσεις πραγματικά μας κάνουν να αρρωσταίνουμε όταν τις διαβάζουμε. Χιλιάδες ροχίνγκια δολοφονούνται καθημερινά. Τα παιδιά τα ίδια. Ε, εθνοκάθαρση είναι αυτό, γενοκτονία. Το 2017 διεξάγεται τέτοια εθνοκτονία και λυπάμαι που κάποιοι συνάδελφοι ακόμα και αυτό το αμφισβητούν. Και οι διεθνεί οργανώσει δεν μπορούν να φτάσουν εκεί. Είναι παγιδευμένοι οι Ροχίνγκια σαν ποντίκια μέσα στη φάκα. Τι θα γίνει, θα ασχοληθεί κάποιο. Και κάθεται μια κυρία εκεί που είναι και βραβευθήσα με βραβείο Νόμπελ Ειρήνη και παρατηρεί. Και είναι και βραβευθήσα και με το βραβείο το δικό μας, το Ζαχάροφ. Καλά είναι να λαμβάνει τίτλου και βραβεία, αλλά πού είναι τα έργα, πού είναι η προστασία των ανθρώπων. Δεν μπορούμε ω Ευρώπη να παραμείνουμε παρατηρητέ. Θα πρέπει να ασκήσουμε την επιρροή μα στον κόσμο για να πιέσουμε και να φροντίσουμε από κοινού να σταματήσουν ε, οι διώξει των Ροχίνγκια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Τζέν Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Και εγώ μιλώ ω πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία για την Νότια Ασία που καλύπτει και τον Μπαγκλαντέ ε, και όπου στο παρελθόν επισκεφθήκαμε του καταβλισμού Ροχίνγκια. Ε, ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, χρηματοδότηση υποστηρίζοντα του Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντέ, του πρόσφυγε που βρίσκονται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα βάζει 3 ε, εκατομμύρια από το Ταμείο ΕΚΟ και ρωτούμε πώς ακριβώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα, δεδομένου ότι καλύπτει και την Μιανμάρ και όπως μόλις ακούσαμε δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε για τον ΟΗΕ ούτε ε, για τις διεθνείς ΜΚΟ ε, στην περιοχή των Ροχίνγκια εντός Μιανμάρ. Ε, πρέπει ε, λοιπόν να έχουμε ενεργή και δραστήρια διπλωματία εντός της περιοχής με τις δύο μεγάλες αυτές ε, δυνάμεις γιατί είναι κάτι που συνεχίζεται. Ο, κόσμος πρέπει να μπορέσει να επιστρέψει στα σπίτια του με αξιοπρέπεια και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο την Αγξανξουκή αλλά τους στρατηγούς και την στρατιωτική τους ισχύ επίσης. Ας μην τους αφήσουμε σε ησυχία. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτ. Και τώρα ο κύριος Ιγνάτσιο Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τραγωδία που πλήττει τον λαό των Οργίνγκια είναι μια πάνθρωπη τραγωδία. Ε, ήδη έχουμε μιλήσει για αυτό τον λαό που πολύ συχνά έχει χτυπηθεί από τον Ιούλιο του 2016 και φέτος το Μάρτιο ξανά άλλο ψήφισμα ψηφίσαμε. Δυστυχώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σύμφωνα με την ΥΠΑ Τερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 300.000 ε, Ροήνγκια προσπαθούν να φύγουν προς τον Μπαγκλαντές για να ξεφύγουν από τις θανατώσεις και τις δολοφονίες, ενώ οι, ε, από φωτογραφίες δείχνουν τεράστιες καταστροφές. Δείχνουμε για έναν ολόκληρο λαό από το 1992 δεν έχει ηθαγένεια, είναι απάτρις. Ε, ε, ε, και μάλιστα έχει ναρκοθετηθεί ολόκληρη η περιοχή για να μην μπορούν να επιστρέψουν ποτέ αυτοί οι ε, πρόσφυγες. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να αποσύρουμε το βραβείο Ζαχάροφ, να ακυρώσουμε την αντιπροσωπεία της ΣΥΝΤΑ που θα πάει την επόμενη εβδομάδα. Υποτίθεται γιατί είναι τρελό να μιλάμε για εμπόριο ενώπιον μιας τέτοιας τραγικής κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοράου. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, ακούσαμε, συνεχίζεται η συζήτηση για τους Ροχίνγκια και στο παρελθόν είχαμε επιληφθεί, αλλά θα πρέπει να καταδικάσουμε και να στυλτεύσουμε αυτή την κλιμάκωση της βίας. Αλλά η απλή καταδίκη δεν βοηθά. Το αντίθετο, είχαμε όξυνση της κατάστασης και ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Πάνω από 300.000 ροχίνγκια εξορίστηκαν, αυτά στον Πακλαντές και μάλιστα ναρκοθετήθηκαν τα σύνορα από τη Μιαμάρ για να μην μπορέσουν να επιστρέψουν. Θα πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένες κυρώσεις και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα για να επιβάλλουν κυρώσεις στην κυβέρνηση Τη Μιαμάρ και επίσης άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τι να κάνει και το Μπάγκλαντε. είναι πολύ εκρηκτική κατάσταση και εκεί. Πρέπει να υποδεχθεί εκατοντάδε χιλιάδε πρόσφυγες Ροχίνγκια. Και είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τις δράσεις της κυρίας Σαξουκή, βραβευτή σας με Νόμπελ Ειρήνης, αλλά ο βασικός υπέτειος και αυτούργος αυτών των θηριοειδών είναι ο στρατός, μην το ξεχνάμε. Καμ. Χαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι φρικαλαιότητες απέναντι στην κοινότητα Ροχίνγκια θα πρέπει να σταματήσουν. Χαιρετίζω το σημερινό ψήφισμα, γιατί η επονίδη στη συμπεριφορά της Άγξαν Σουκή οφείλεται στο φόβο ότι αν υπεράσπιζε τους Ροχίνγκια θα προκαλούσε την ε, ε, θυμωμένη, οργισμένη αντίδραση του στρατού. Αλλά είναι ντροπή να μένουμε απλοί θεατές ε, μία γενοκτονία. Και σίγουρα ε, δεν ήταν ε, ε, σωστή αντίδραση ούτε Βρεβευθείς με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ούτε οποιοδήποτε δημοκρατικού ηγέτη. Θα πρέπει να φροντίσουμε για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να ασκήσουμε και επίση και στην Κίνα, που έχει κάποια επιρροή στο στρατό της Μιανμάρ. Και όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Δέσμον Τούτου, μια χώρα που δεν είναι συμφιλωμένη, δεν είναι σε ειρήνη με τον εαυτό της, δεν μπορεί να και που δεν μπορεί να προστατεύσει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των λαών που διαβίωσαν αυτή δεν είναι ελεύθερη χώρα. Κυρία Ανσαξουκή, στρεφόμαστε προς εσάς για να βοηθήσετε τους Ροχίνγκια. Σας παρακαλούμε θερμά και για τους Ροχίνγκια και για την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση. Δεν είναι πρώτη φορά που η μουσουλμανική μειονότητα των Ροίνγκια στη Μιαμάρ υπόκειται σε βία. Ε, περιορισμό ε, των πάντων, απειλέ στη ζωή και στην ασφάλεια, άρνηση του δικαιώματο στην υγεία και στην παιδεία και περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο ειδικό ε, ε, εισηγητή του ΙΟΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλά για ήδη ένα εκατομμύριο 250.000 πρόσφυγες που, ε, Ροχίνγκια που έχουν φύγει προς τον Μπαγκλαντέ. η ηγέτης τη της Μιανμάρα απορρίπτει τις ε, κατηγορίες καταστολής και ή εθνοκάθαρσης απέναντι, ε, εναντίον μάλλον των Ροχίνγκια. Και μάλιστα λέει ότι πρόκειται για ψευδείς ειδήσει. Απέναντι σε αυτή την κυρία θα πρέπει να στραφούμε ώστε να βρεθεί μια λύση ειρηνική που θα λαμβάνει υπόψη την αξιοπρέπεια και τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καπούτο και τώρα τέλος η Αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Μιανμάρ έχει περάσει σχεδόν μισό αιώνα στρατιωτικού νόμου και απομόνωσης. Ορισμένοι αναφερθήκατε στην ιστορία και στο παρόν ακόμα της χώρας, ότι δηλαδή ε, κυριαρχεί ο στρατός και μάλλον έχετε δίκιο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα γεγονότα τα, των τελευταίων ημερών ε, ταυτόχρονα με την ιστορία. Έχει κάνει ωστόσο εντυπωσιακέ αλλαγέ αυτή η χώρα τα τελευταία χρόνια και ωστόσο δεν έχει ολοκληρώσει το δρόμο προς την ε, δημοκρατία. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τις επιθέσεις της 25ης ε, ε, της, 25ης 8 καθώς και όλες τις υπόλοιπες επιθέσεις που έγιναν στο κρατήδιο Ραχίν και πιστεύουμε ότι οι δράστες θα πρέπει να ε, δικαστούν. Και να πω ξεκάθαρα, όπως το έχουμε ήδη δηλώσει, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ανησυχούμε για τις υπερβολές που έγιναν από τις δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρα. Αυτό οδήγησε σε μαζική ροή προσφύγων προς τον Μπαγκλαντές είναι μια από τις πιο φρικτές προσφυγικές κρίσεις ε, των καιρών μας. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε δύο άμεσες προτεραιότητες και με χαρά είδα που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησε το θέμα χθες το βράδυ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε παρόμοιες προτεραιότητες με αυτές που θα σας αναφέρω και εγώ ε, σε λίγο. Πρώτη άμεση ε, προτεραιότητα να πάψουν οι εχθροπραξίες, η βία να σταματήσει, να υπάρξει αποκλιμάκωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά από όλους, αλλά είναι σαφές ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ε, φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για να περιορίσουν τις βίες ενέργειες απέναντι εναντίον μάλλον άοπλων πολιτών. Έπειτα θα πρέπει να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε όσου τη χρειάζονται. Ε, και μάλιστα πηγόντω. Εδώ πρέπει να παίξουμε το ρόλο μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πράττουμε με αξιμίωτο τρόπο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Στυλιανίδη για την αφοσίωση την εργασία του που αποδεικνύεται ουσιαστική αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίπτωση. 350.000 ευάλωτοι άνθρωποι υπάρχουν στο Ραχήν. Ε, πρέπει γρήγορα να φτάσει εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια και για πολλούς αυτό σημαίνει είναι ζήτημα ζωή και θανάτου. Ο συνάδελφος Τηλιανλίδης και εγώ συνεργαζόμαστε πολύ στενά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και χτε, μετά από δική μας επιμονή και πολύ διπλωματική δουλειά η κυβέρνηση επικοινώνησε με το Διεθνή ε, Ερυθρό Σταυρό και είπε ότι θα το επιτρέψει να μπει στη χώρα και να πάρει 30.000 κόσμο, να βοηθήσει 30.000 κόσμο. Ε, είναι μόνο η αρχή και ελπίζουμε πως θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια γιατί οι αρχές του Μπαγκλαντές έχουν καλωσορίσει πολλούς ε, ε, πρόσφυγες και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει μόνο να επενέσει αλλά και να στηρίξει τις προσπάθειες αυτής της χώρας. Και ως άμεση απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αυξήσει τη στήριξή της προς τον Μπαγκλαντές με ακόμα 3 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον των 12 ε, που ήδη προδίνονται στην Μιανμάρ και στον Μπαγκλαντές μαζί. Αυτές είναι οι δύο άμεσες προτεραιότητες, να σταματήσει η βία και να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά μετά έχουμε και άλλο ένα σημαντικό έργο, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε με όλους όσοι εμπλέκονται για να εξευρεθεί μια μόνιμη ειρήνη ε, στην Μιανμάρ, να εξετάσουμε και να λύσουμε το μόνιμο θέμα των Ρογινγκιά. Όπως ξέρετε δεν είναι η πρώτη φορά, ε, τώρα είναι μια οξία κρίση και πέρα από αυτό πρέπει να εργαστούμε για το πολιτικό σκέλος. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι μία από τις, ε, ε, ε, τα αίτια της αστάθειας στην περιοχή είναι το στάτους των Ροχίνγκια. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πάντοτε το ζητούσαμε, ανέκαθεν το ζητούσαμε στο πολιτικό διάλογο με τη Μιαμάρ στα διάρκεια των ετών και στα επαφέ υψηλού επίπεδου, αλλά και στο διάλογο Ευρωπαϊκή Ένωση Μιαμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελευταίο Μάρτιο, τον περισμένο Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο συζήτησε για αυτό το θέμα και υπάρχει και πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συστάσεις ε, της ε, ε, για την χώρα αυτή από τον Κόφι Ανάν είναι η αναφορά μας. Η κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει υποσχεθεί να προωθήσει αυτά τα θέματα και εγώ συζήτησα προσωπικά με την Άγξαν Ξουκή αυτά τα θέματα στην επίσκεψή της στις Βρυξέλλες πριν από λίγους μήνες. Ε, εξάλληψη των διακρίσεων, ελάφρυνση της στόχιας, εξασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίση πρόσβαση στην παιδεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και πρόθεση της εμπιστοσύνης και της συμφιλίωσης. Ο χρόνος εφαρμογής της έκθεσης Σανάν είναι τώρα, γιατί βλέπουμε τι αντιμετωπίζει ο λαός του Ράκιν και δεν μπορεί να περιμένουμε άλλο. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την εφαρμογή αυτών των συστάσεων με κάθε τρόπο. Η κυβέρνηση της ε, Μιανμάρ θα πρέπει επίσης να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ και να την ενισχύσει καθώς και με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ, αλλά και με ε, την, την ε, ανεξάρτητη αποστολή ανέβρεσης στοιχείων και αυτό το συζητήσαμε με την Άξαν Σουκή και όλα αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την κυβέρνηση της Μιανμάρ θα, εξε, θα εξεταστούν από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως από την αντιπροσωπεία μας εκεί ε, εξετάζονται καθημερινά και συζητώνται καθημερινά. Με τον ΟΗΕ συνεργαζόμαστε, προσωπικέ επαφές έχω με τον Γενικό Γραμματέα Κουτέρης και με τους συναδέλφους ε, σε ολόκληρο τον κόσμο για αυτό το θέμα και θα χρησιμοποιήσουμε τη Γενική Γραμματεία, ε, συγγνώμη, την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την Υπουργική Εβδομάδα ώστε να το συζητήσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι η διεθνή κοινότητα θα μείνει ενωμένη. Η πορεία της Μιανμάρ προς τη δημοκρατία αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς στον κόσμο και για μένα προσωπικά και πιθανότητα και πολλούς για εσάς εδώ σε αυτή την αίθουσα. Η ευθύνη της ηγεσία της χώρας ε, της πολιτικής αλλά και της στρατηγικής ε, ε, ηγεσία είναι τεράστια. Ακριβώς επειδή